την κυρία Πλάμπ για την εκλογή της και θα μπορούσε να τα διαβιβάσει αυτά τα συγχαρητήρια ο κύριος Σφόμποντα. Επίσης, η, η εντολή της κυρίας Λάγγεν έχει εγκριθεί ομόφωνα από την αρμόδια επιτροπή και από την 17η Μαρτίου θεωρείται ότι έχει ελεγχθεί η εντολή της και έχει τα πλήρη δικαιώματα οποιοδήποτε βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν αντίρρησεις, δεν είναι ούτως. Επομένως, έχει επικυρωθεί και από την Ολομέλεια ο έλεγχος της εντολής. Η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων